Και αυτή είναι απλά η αρχή. Ευχαριστώ κυρία Καϊλή. Το τελευταίο μου σχόλιο είναι ότι ε, ε, θα έχουμε μια πολύ ωραία δεξίωση στη συνέχεια να μπορούμε να συζητήσουμε άνθρωπο προς άνθρωπο, πρόσωπο με πρόσωπο και άμα θέλετε να μιλήσετε με κάποιον πάτε παρακάτω έτσι. Μείνετε πάντως για τη δεξίωση γιατί είναι ένα σημαντικό σημείο της συζήτησης στην πραγματικότητα. Να πω επειδή κάποιοι είπαν, αναφέρθηκαν στο Tommy X, ε, είχαμε πολλές πληροφορίες και σήμερα, ε, ευχάριστος πονοκέφαλος αυτός, θέλω να είμαστε ανοιχτοί, διαφανείς, είναι καλό ότι μπορείς να έρθει ο κ. Μέτσιγκερ να είναι ανοιχτό, να διαφανείς πριν τη δημοσίευση του εγγράφου. Αυτό είναι πραγματικά καλό. όλες οι παρουσιάσεις ε, και από τις θρησκευτικέ ε, οργανώσεις ε, και από τις ανθρωπιστικές οργανώσεις ήταν εξαιρετικές. Είναι μάλλον το τελευταίο μου ανοιχτό σεμινάριο για τον διάλογο στα πλαίσια του άρθρου 17. πραγματικά εντυπωσιάζομαι που βρίσκονται τόσοι άνθρωποι σήμερα στην αίθουσα, διότι αυτό το θέμα θα μας απασχολήσει στο μέλλον. Θα είναι το θέμα του μέλλοντος και το πιο σημαντικό είναι η κριτική σκέψη. Το κάνω και εγώ. Πιστεύω ότι και στην πολιτική ζωή δεν το κάνουμε αρκετά αυτό. Δεν έχουμε τον χώρο, δεν έχουμε τον χρόνο, ε, δεν υπάρχει ο χώρος που να μην, μας, που να μην εισβάλλει τεχνολογία. Γι' αυτό συνήθω πάω σε κάποιο λιβάδι με ένα ε, ε σκύλο και είναι κάτι που επιτρέπει στο μυαλό μου να χαλαρώσει και να σκεφτεί χωρίς ε, την συνεχή επαφή με την τεχνολογία. Και ως πολιτικοί θύνοντες ε, έχουμε απέναντί μας πιο ε, έτσι ανυπόμονους πολίτες. Μας στέλνουν κατευθείαν στο Twitter, δεν μας στέλνουν επιστολές ε, και είναι και live τώρα η ε, συγκεκριμένη εκδήλωση. Το Facebook, τα SMS που λαμβάνουμε θέλουν απάντηση αμέσως και πρέπει οι πολιτικοί θύνοντες να ξαναπάρουν τον έλεγχο και μπορεί να μας βοηθήσετε ίσως και προς την κατεύθυνση αυτή για να παίρνουμε και καλύτερες αποφάσεις ε, υπέρ των πολιτών. Οι συνάδελφοι εδώ θεωρούν ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι για καλό, αλλά πάντα υπάρχουν σε όλες τις εξελίξεις του ανθρωπότητας υπάρχουν και αρνητικά στοιχεία. Αυτό που δεν μπορούμε να δεχτούμε είναι ότι έχουμε χάσει τον έλεγχο. Αυτό δεν μπορούμε να το κάνουμε ε, και δεν πρέπει. Γι' αυτό λοιπόν είναι σημαντικό αυτό το σεμινάριο όπου έχουμε εδώ ε, εκπροσώπους θρησκευτικών δόγματων, ε, ανθρωπιστικών οργανώσεων και είναι πολύ θετικό ότι είμαστε τόσοι εδώ ε, και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο βεβαίως που συμμετείχαν στο διάλογο καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Ε, θα ήθελα να κάνω κάποια συμπερασματικά, κάποιες σημαντικές παρατηρήσεις για το διάλογο αυτό το οποίο προείσταμε εδώ και δυόμιση χρόνια. Ο κ. Σταγιάννη λυπάται που δεν μπορούσε να έρθει σήμερα. Ήθελε να είναι εδώ κατά τα τελικά σχόλια. Πιστεύω ότι ο διάλογο αυτό ήταν αναζωογονητικό. Τα τελευταία αυτά δυόμιση χρόνια έμαθα πολλά. Έμαθα επίση ότι πρέπει να κάνουμε περισσότερα και καλύτερα. Θέλω να ευχαριστήσω λοιπόν όλου όσους συνεισέφεραν στα συμπεράσματα αυτά. Ε, τα είπα και στο Προεδρείο, θα τα πω μάλλον πριν τι επόμενε εκλογέ, διότι αυτό ο διάλογο θα πρέπει να διευρυνθεί ε, να μην συζητάμε μόνο μεταξύ μας, να φτάσει και σε επιτροπές όπου σήμερα αποδείξαμε ότι μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο. Είναι για το ευρύτερο καλό. Για όσους με υποστήριξαν στο έργο μου από τις οργανώσεις εδώ, από τις εκκλησίες, σας ευχαριστώ όλους για την υπομονή σας, διότι δεν είχα και επαρκή γνώση ενδεχομένως αρχικά. Ε, αναγνωρίσατε τη δουλειά που προσπάθησα να κάνω στο όνομά σας. Θέλω να ευχαριστήσω τον Φέργκου Σοχάρα, ο οποίος είναι εδώ πίσω μου σιωπηλά, ε, χάρηκα που συνεργάστηκα μαζί του και με το γραφείο του και τον Τζόρτζο Χέι, τον, βοηθό μου, που είναι συνήθω κάπου στο βάθο, αλλά κάνει πραγματικά εξαιρετική δουλειά. Θέλω πραγματικά να χειροκροτήσετε όλους όσους ε, βοήθησαν για να συμβεί αυτό. Να ευχαριστώ την κυρία Καϊλή τους συναδέλφους ε, ευρωβουλευτές, διότι είμαστε τόσο καλοί, είναι αυτοί που μας υποστηρίζουν, μην το ξεχνάμε αυτό. Έχει γίνει πολύ καλή δουλειά ε, από τους υπαλλήλους και στο Κοινοβούλιο και στην Κομισιόν. Όπως είπα, ε, αυτό είναι η τελευταία. Η τελευταία συνάντηση, εξού και δεξίωση, εξού και πάρτι αν θέλετε μετά. Ανταλλάξτε απόψεις, πληροφορίες, ε, κάρτες. Εγώ δεν χάνω την εμπιστοσύνη μου και την πίστη μου στην ανθρωπότητα, επειδή όμως έχω τέσσερα παιδιά Νομίζω ότι οι γονείς έχουν την αίσθηση ότι χάνουν τον έλεγχο, όχι με την κακή έννοια των παιδιών, αλλά υπάρχουν πάρα πολλές επιρροές εξωτερικές και το νιώθουν αυτό οι γονεί ότι δεν ελέγχουν. Ο, ο μικρότερος γιος μου θα είναι 18 σύντομα και χαίρομαι που δεν είναι 8, γιατί δεν νομίζω ότι θα μπορούσα να αντιμετωπίσω όλα αυτά που έρχονται πάνω μα. Εν πάση περιπτώσει, η σημερινή μα εκδήλωση μας δώσει, θα μα δώσει ενδεχομένω κατευθύνσεις γραμμές και τον Απρίλιο να μένουμε και το έγγραφο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Νομίζω ότι ήταν προνομιακό για μα ότι λάβαμε κάποια πρώτα στοιχεία αυτού σήμερα και βεβαίω ήταν ε, πραγματικά τιμή για μα που είχαμε πυρογνώμονε και στα δύο πάνελ σήμερα ε, και θα πρέπει νομίζω όσους ήρθαν να μιλήσουν εδώ να τους ε, ευχαριστήσουμε και να του χειροκροτήσουμε. Τους ευχαριστώ όλους και πάμε τώρα όλοι στη δεξίωση. σα ευχαριστώ πολύ.